Okay, colleagues, we can uh, welcome back to the second day of our committee. Um, Συνάδελφοι, καλημέρα σας. Είχαμε τη συνεδρίαση των συντονιστών από τις 9 και ορισμένοι θερμινοί είναι εδώ από το πρωί, οπότε έχει έρθει η ώρα να συνεχίσουμε. Σήμερα θα αρχίσουμε με το σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης, χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα όπως ξέρετε, τον Ιούλιο θα γίνει διάσκεψη στην Αντίσα Μπέμπα, όπου η παγκοσμία κοινότητα θα δει πώς θα χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη για τα επόμενα 15 χρόνια μετά το 2015 και αυτό θα έρθει να προσθεθεί και στη διάσκεψη των ΗΠΑ το Σεπτέμβριο. Σήμερα το απόγευμα, μετά την συζήτησή μας για τα ορυκτά, θα έχουμε μια ακρόαση. Ο κύριος ε, Περέιρα θα σας πει περισσότερα για αυτή, αλλά θα ασχοληθούμε με ένα από τα σημαντικότερα θέματα που έχουμε να... ως Επιτροπή. Πριν από δύο περίπου εβδομάδες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πρόταση Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης και είχαμε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας ως απάντηση της ανακοίνωσης αυτής της Κομισιόν στοχεύουμε να ψηφίσουμε αυτή την έκθεση πριν το επίσημο Συμβούλιο στα τέλη Μαΐου, έτσι ώστε να επηρεάσουμε τα αποτελέσματα της συνεδρίας του Συμβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς καμία καθυστέρηση, θα δώσω αμέσω το λόγο στον κύριο Σίλβα Περαίρα, Πέντρο, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να πω πως καλωσορίζω την ευκαιρία για να έχουμε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Όπως είπατε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ πρόσφατα παρουσίασε μια ανακοίνωση σχετικά με την παγκόσμια συνεργασία για την απαλληφή της φτώχειας και την βιώσιμη ανάπτυξη μετά το 2015. Αυτή τη στιγμή επεξεργάζομαι το σχέδιο έκθεσης. Θα σταλεί σύντομα για μετάφραση. Έχει γίνει όμως ήδη μια πρώτη συνάντηση με τους κοιόδης εισηγητές και Διοργανώσαμε μια συνάντηση με μη κυβερνητικέ οργανώσεις στι αρχές Φεβρουαρίου. Και όπως είπατε πολύ σωστά και εσεί, σήμερα το απόγευμα θα έχουμε μια επίσημη δημόσια ακρόαση για το θέμα αυτό. Όπου θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Επίτροπο Μίμητσα και άλλους ενδιαφερόμενους μη κυβερνητικέ οργανώσει, αλλά και φορείς του ιδιωτικού τομέα και διεθνεί οργανισμού. Σχετικά τώρα με το χρονοδιάγραμμα της έκθεσης του Κοινοβουλίου, να σας πω ότι η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι η 23η Μαρτίου. Ψηφοφορία στην Επιτροπή 20 Φεβρουαρίου, 20 Μαρτίου και στην Ολομέλεια το Μάιο. Για να προλάβουμε τη συνεδρίαση του Συμβουλίου και το συνεδρίο της Αντίσα Μπέμπα τον Ιούλιο. Μας μένουν 20 εβδομάδες μέχρι τη διάσκεψη στην Αντίσα η οποία φυσικά διάσκεψη είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι το αποτέλεσμά της αναμένεται να σκιαγραφίσει πώς ο κόσμος θα αντιμετωπίσει τους ε, αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική η έκθεση αυτή, διότι θα δημιουργήσει ένα προηγούμενο για τις επόμενες διασκέψεις στη Νέα Υόρκη και το Δεκέμβριο για, στο Παρίσι για το κλίμα. Είναι πάρα πολύ σημαντική λοιπόν αυτή η προπαρασκευαστική περίοδος πριν την Αντισαμπέμπα. Θα χρειαστεί να εγκρίνουμε ένα σχέδιο δράσης για να έχουμε ένα λειτουργικό επιχειρησιακό σχέδιο και όπως είπα έχουμε 20 εβδομάδες για να έρθουμε σε μια πολιτική συνεννόηση. Θα συζητηθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας, οι ανάγκες χρηματοδότησης που ανέρχονται περίπου σε 3-3 εκατομμύρια δολάρια να έτος και μας λείπουν τα 2,5 από αυτά. Χρειάζεται λοιπόν δράση για να κινητοποιήσουμε πόρους. Χρειαζόμαστε λοιπόν καλή συνεργασία και ιδιαίτερα να προωθήσουμε τη συνεργασία και με τα Ηνωμένα Έθνη έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε μια παγκόσμια προσπάθεια και μια σημαντική συνεργασία με όλους τους φορείς. Και πιστεύω πως, όπως και εσείς φαντάζομαι θα συμφωνείτε μαζί μου, ότι όλες οι δυνατότητες συνεργασίας πρέπει να εξαντληθούν και καθώς και όλες οι ικανότητες επίσης. Έχουν αλλάξει σημαντικά τα δεδομένα τα τελευταία 15 χρόνια και πρέπει να ληφθεί υπόψη και η κατάσταση στις αναδυόμενες οικονομίες Έχει αλλάξει επίσης και η κατάσταση όσον αφορά τα εισοδήματα στις ε, χώρες με μικρά και μεσαία εισοδήματα. Γι' αυτό λοιπόν είναι και λογικό να αναμένουμε από τις χώρες εταίρους μας διαφορετικού είδους δέσμευση για το μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια παραμένει ο μεγαλύτερος δωρητής αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο και είναι πάρα πολύ σημαντική λοιπόν η συνδρομή μας. Και αναμένουμε αυτή η αναπτυξιακή βοήθεια να συνεχίσει να είναι υψηλή και στο μέλλον. Πιστεύω λοιπόν πως η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να τύχει της υποστήριξής μας, πρέπει να αναγνωρίσουμε την πολιτική της θέληση, διότι αναφέρεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να εξαντλήσει τις αρμοδιότητές της και αυτό θεωρώ πως είναι ένα πάρα πολύ καλό σημάδι πολιτικής δέσμευσης. Φυσικά πρέπει να συζητηθούν πολλά πολιτικής φυσιοζητήματα πριν αρχίσουμε την, τις διαβουλεύσεις μας και καταρχάς θα ήθελα να πω ότι η δική μου εκτίμηση είναι ότι υπάρχει έλλειψη δέσμευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι ανησυχητικό και αρνητικό πολιτικά και δημιουργεί επισφάλεια για το μέλλον της διαδικασίας. Ορισμένες μη κυβερνητικέ οργανώσεις επίσης αναφέρονται σε έλλειψη ε, φιλοδοξίας. Εγώ θα έλεγα πως είναι περισσότερο έλλειψη δέσμευσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει πως θα έπρεπε να γίνει εκ νέου δέσμευση για τον στόχο του 0,7% όμως, το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη του στόχου αυτού πρέπει να εξαρτάται από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με τους υπόλοιπους εταίρους μας παγκοσμίω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στήριξε τον στόχο τη Γενικής Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών, όμως υπάρχει και ένας στόχος για το χρονοδιάγραμμα και να σας πω ότι υπήρχε ήδη ένα χρονοδιάγραμμα και από εμάς. Γι' αυτό λοιπόν, εάν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι αξιόπιστη, πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω. Πέρα από το ότι δεσμεύεται για τους στόχους. Πρέπει να είναι έτοιμη να παρουσιάσει ένα χρονοδιάγραμμα και έναν εποπτικό μηχανισμό ο οποίος θα ελέγχει την τήρηση του χρονοδιαγράμματος αυτού. Και πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη ότι χρειάζεται ηγετική παρουσία στη διάσκεψη της Αντισαμπέμπα. Διαφορετικά κινδυνεύει η εξοπιστία μας. Και αυτό θα υπονομεύσει τις πιθανότητες να οδηγηθούμε σε καλά αποτελέσματα στην Αντισαμπέμπα. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι υπάρχει έλλειψη δέσμευσης. Επίσης υπάρχει το ζήτημα της χρηματικής υποστήριξης, οικονομικής υποστήριξης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Γιατί πρέπει όλες οι χώρες με χαμηλά... Όλες οι χώρες ανεξαρτήτως εισοδήματος να σέβονται τον, το στόχο του 0,7 100. Αλλά πιστεύω πως θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε πέρα από αυτό, να έχουμε ένα 0,2% έστω. Και θα έπρεπε να το εξετάσουμε. Φυσικά, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αυτή τη στιγμή συζητιέται το τι είναι η επίσημη βοήθεια. Και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση, διότι εμείς επιθυμούμε οι στόχοι μας να είναι ουσιαστικοί και δεν θέλουμε έναν καινούριο ορισμό, ο οποίος όμως να περιέχει στην ουσία τα ίδια πράγματα και τους ίδιους πόρους. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι συζητήσεις που γίνονται για τους ορισμούς, καθώς και για τις επιπρόσθετες λεπτομέρειες. Τη χρηματοδότηση στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής, για παράδειγμα. Έπειτα, δεύτερο πολιτικό ζήτημα είναι η εγχώρη πόροι Και εδώ να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ σωστά τόνισε ότι πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι οι εγχώροι πόροι και αυτό απαιτεί ένα σωστό σύστημα φορολόγησης. Και πιστεύω πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να προσπαθήσει να διασφαλιστεί μία σωστή διεθνή συνεργασία για τη φορολόγηση, διότι το φορολογικό σύστημα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεών μας. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τις νέες πηγές χρηματοδότησης και για το πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. χρηματοπιστωτικούς φόρους, για παράδειγμα, περιβαλλοντικούς φόρους. Πώς μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις νέες πηγές για την ανάπτυξη. Και αυτό είναι το δεύτερο λοιπόν πολιτικό σχόλιο. Και επιπλέον θα ήθελα να πω κάτι για τον ιδιωτικό τομέα. Φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμπεριληφθεί ο ιδιωτικός τομέας, διότι υπάρχει τεράστιο δυναμικό εκεί. Αυτό όμως σημαίνει και πως ε, πρέπει να συζητηθούν οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα εναρμονιστεί ο ιδιωτικό τομέας με τους ε, στόχους για την αηφόρο ανάπτυξη. Πώς θα γίνει αυτό δηλαδή, ποια χρηματοδοτικά μέσα χρειάζονται. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να συμπεριληφθεί και αυτό στις πολιτικές μας συζητήσεις. Και τέλος, διαφάνεια, λογοδοσία και καταπολέμηση της διαφθοράς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν συζητούμε για αυτά να είμαστε σίγουροι πως τα χρήματα πηγαίνουν στο σωστό μέρος και στο σωστό σκοπό. Και φυσικά πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η λογοδοσία. Και πρέπει αυτή να είναι και η πολιτική τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν γέννη. Να δοθεί έμφαση λοιπόν στο ζήτημα αυτό. Αυτά ήταν τα πολιτικά σχόλια που ήθελα να κάνω τώρα στην αρχή. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να συζητήσουμε, παγκόσμια διακυβέρνηση για παράδειγμα, όμως πιστεύω πως ε, είναι καλή αφορμή αυτά τα λίγα σχόλια για να αρχίσει η συζήτηση και ανυπομονώ να συζητήσω λοιπόν μαζί σας, να ανταλλάξουμε απόψεις, ιδιαίτερα με τους σκιώδεις εισηγητές, έτσι ώστε η έκθεση να είναι όσο το δυνατόν περιεκτικότερη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω τον Πολυρούμπικ ε, πρώτα και τους κοιόδης όλους, μας περιπτώσει. Ναι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την πολύ καλή συζήτηση σε σχέση με τούτη την έκθεση. Θα συνεχίσω λοιπόν στα γερμανικά, στη μητρική μου γλώσσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα τον Σίλβιο Περέιρα, διότι πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλου μα πιστεύω να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι για την αηφορία και τη βιωσιμότητα και είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία ανάμεσα στη, στα κράτη-μέλη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και του διεθνεί οργανισμού. Και φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο εδώ. Και μάλιστα έχουμε και τους 17 στόχους που έχουν τεθεί για εν ώψη της διάσκεψης στη Νέα Υόρκη και πρέπει να δούμε βήμα-βήμα πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες για τον καθένα από αυτούς. Ε, ενέργεια, λοιπόν, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το κυριότερο, διότι χωρίς ενέργεια δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η ενέργεια, λοιπόν, είναι ιδιαίτερα σημαντική, ιδιαίτερα στον, ε, στην Ήπεθρο και στις αγροτικές περιοχές. Και πιστεύω επίσης πως ε, πάρα πολύ σημαντικό για την υγεία είναι το καθαρό νερό. Αυτές είναι οι βάσεις έτσι ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και να διασφαλιστεί και η αηφορία της. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και αυτό χρειάζεται μία διατομιακή συνεργασία. Επίσης η συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική προϋπόθεση. Το χρήμα δεν θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Αντίθετα, Πιστεύω πως στο επίκεντρο πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Να σας αναφέρω ενδεικτικά ότι 1,3 δισεκατομμύρια ε, άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν ηλεκτρισμό. 2,6 δισεκατομμύρια μαγειρεύουν ακόμα χρησιμοποιώντας βιομάζα για πηγή ενέργειας. Χρειάζεται λοιπόν μία σύγχρονη πρόσβαση σε ενέργεια για όλους. Μπορούμε να δούμε επίσης την περίπτωση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στοιχείων ε, στην Αφρική ή εγκαταστάσεις ε, επεξεργασίας βιομάζας στην Ασία, στον Παγκλαντές για παράδειγμα. Μπορούμε να δούμε με αυτά τα προγράμματα ότι υπάρχει δυναμικό για περισσότερη ανάπτυξη. Και εδώ να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι χώρες που βρίσκονται κοντά στον Ισημερινό, διότι έχουν μεγάλα ενεργειακά αποθέματα ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Πιστεύω επίσης ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο να γίνεται μεταφορά πόρων από ε, τις αναπτυγμένες, τις αναπτυσσόμενες χώρες. Πρέπει να δούμε και πέρα από αυτό και σε αυτό θα παίξει ρόλο και η Επιτροπή Προϋπολογισμού. Πρέπει να δούμε λοιπόν την απόδοση και το αποτέλεσμα της ε, αποδοτικής χρήσης των κονδυλίων αυτών. Έτσι ώστε να αποφύγουμε διάφορες περιπτώσεις φοροαποφυγής ή κοντιλίων τα οποία πηγαίνουν στις αναπτυσσόμενες χώρες ως αναπτυξιακή βοήθεια και καταλήγουν σε διάφορες offshore εταιρείε ή αλλού. Πρέπει λοιπόν να διασφαλιστεί η σωστή χρήση των πόρων. Επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε την υποστήριξη στο σύστημα των μικροπιστώσεων στις ε, στα πλαίσια της αναπτυξιακής βοήθειας. Μικροπιστώσεις ε, θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν, για παράδειγμα, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, το, οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ε, επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμπεριληφθεί και ο ιδιωτικός τομέας, ιδιωτικές επενδύσεις, έτσι ώστε να ενισχυθεί η αναπτυξιακή βοήθεια. Και πιστεύω εδώ πως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο μέλλον και όχι μόνο αυτή, αλλά και το επενδυτικό σχέδιο του ε, Jean-Claude Juncker. Τα περίφημα 315 δισεκατομμύρια. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποια έργα θα μπορούσε να στηρίξει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στις αναπτυσσόμενες ε, χώρες. Είναι πέραν αυτού πάρα πολύ σημαντικό να σταματήσουν, να σταματήσει η παράνομη εκροή πόρων γιατί υπολογίζεται ότι εκατοντάδες δισεκατομμύρια διαφεύγουν κάθε χρόνο. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική η καταπολέμηση της ε, διαφθοράς. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνδράμει λοιπόν στην καταπολέμησή της με τις ε, δομές που ήδη διαθέτει και με την ε, διοικητική και διαρθρωτική βοήθεια. Για την σωστή καταπολέμηση λοιπόν των παράνομων χρηματικών συναλλαγών. Επίσης, ας μην ξεχνάμε πως έχουμε και υπαρκτά προβλήματα, δηλαδή την αύξηση των κονδυλίων από 0,15% σε 0,7%. Ας μην ξεχνάμε πως υπάρχουν χώρες όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία που έχουν οικονομικά προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να δούμε εάν αυτός ο στόχος της αύξησης είναι εφικτός για αυτές τις χώρες. Και πρέπει η διεθνής κοινότητα να αναλογιστεί πώς θα στηριχθούν στο μέλλον περισσότερο Ας πάρουμε ένα παράδειγμα ε, τώρα από την Ασία. Η Νότια Κορέα ήταν λήπτης αναπτυξιακής βοήθειας και την χρησιμοποίησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και πρέπει λοιπόν να ακολουθηθεί το παράδειγμα της και από άλλες χώρες. Και πιστεύω εδώ πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά και να αναζητήσει εταίρους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι για λόγους σαφήνειας θα πρέπει ε, να αντιμετωπίσουμε όλες τις μορφές χρηματοδότησης και ευχαριστώ τον ε, εισηγητή Σίλβα Περέιρα που με το γνωστό του τάλαντο ε, κατάφερε να κάνει μια σωστή εισαγωγή στο θέμα. Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά σαφείς στους διάφορους τρόπους χρηματοδότησης. Πρώτον, ε, υπάρχει η δημόσια παρέμβαση, οι δημόσιες επενδύσεις λοιπόν, για την ε, δημόσια βοήθεια για την ανάπτυξη. <clears throat> Αλλά δεν μπορούμε να ασχοληθούμε και να επικεντρωθούμε αποκλειστικά με αυτή τη μορφή. Αναφέρομαι και στην ιδιωτική χρηματοδότηση ε, οποιαδήποτε κονδύλι ε, φτάνει από τις χώρες μας ε, στην Αφρική ή στις χώρες της Αφρικής ε, δεν είναι απαραίτητα κονδύλια προς την ανάπτυξη. Μπορεί να αναφέρονται και σε άλλες διαδικασίες. Επίσης υπάρχει η ανάμειξη ιδιωτικών και δημοσίων και υπάρχει και η ανταλλαγή. Τι σημαίνει αυτό. Ε, εγώ σου δίνω, ε, εγώ κάνω μια επένδυση, εσύ ε, σαν αντάλλαγμα μου δίνεις το δικαίωμα εκμετάλλευσης, άρα δημιουργούμε μια εταιρική σχέση και αυτό δεν θα πρέπει να το παραβλέψουμε. Αυτή η διαδικασία που υπάρχει σε μερικές αναδυόμενες χώρες θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται βάσει των αρχών των Παρισίων και της δακάρα γιατί ε, πραγματικά θα πρέπει να καλέσουμε τους πολιτικούς μας ταγούς ε, και τους υπευθύνους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Κομισιόν να λάβει υπόψη και αυτά τα στοιχεία. Ε, ε, η φύγη κεφαλαίων, το έχουμε αναφέρει αυτό. Και επίσης η διαγραφή του χρέους ε, και αυτό εκλαμβάνεται ως χρηματοδότηση λαμβάνοντας υπόψη και τα όσα αναφέρει και ο Το θέμα αυτό νομίζω ότι δεν είναι πλέον επίκαιρο γιατί τα χρέη τα περισσότερα είτε έχουν διαγραφεί είτε έχουν ξεχρεωθεί, ξεπληρωθεί. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ε, κονδύλι, το μεγαλύτερο ποσό το οποίο ε, αναφέρεται στην ανάπτυξη είναι αυτό το οποίο παράγεται από τις ίδιες αναπτυσσόμενες χώρες. Δεν θα πρέπει δηλαδή να υποτιμήσουμε την ε, ικανότητα των χωρών να βοηθήσουν στην ανάπτυξή τους συμβάλλοντας με ίδιους πόρους. Επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει οι πολιτικοί μας ε, υπεύθυνοι ε, να κληθούν, γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε ε, τέτοια αρμοδιότητα, θα πρέπει όμως να βοηθήσουμε τους αντιπροσώπους μας στην Αντίσα Μπέπα, θα πρέπει να καλέσουμε τους πολιτικούς υπεύθυνους και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να λάβουν υπόψη τις εξελίξεις. Το 2002, να δούμε τι έχει αλλάξει σε σχέση με το Μοντερέι. Ε, είχα πει και στους συντονιστές ε, ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν αλλάξει σε σχέση με το Μοντερέι. Ένα εξ αυτών, ουσιώδες, είναι ότι η Αφρική πλέον έχει γυρίσει σελίδα όσον αφορά το χρέος. Αυτό είναι μια απολύτως καινούρια πρωτόγνωρη κατάσταση. Και δεν το περιμέναμε ότι θα συμβεί αυτό έχει αλλάξει και κάτι άλλο. Ε, η τύχη των αναδειωμένων χωρών. Αυτή η ικανότητα, και το λέω και το ξαναλέω και το επαναλαμβάνω, η ικανότητα που έχουν ε, να δημιουργήσουν, να παράξουν ε, πόρους και δυνατότητες και επομένως εμείς θα πρέπει να είμαστε εκεί μέσω τεχνογνωσίας να τις βοηθήσουμε. Ε, και ε, θα πρέπει να σταματήσει πλέον αυτό το παιχνίδι όπου εμείς στρεφόμενοι προς αυτές τις χώρες λέμε «Α, δεν θα αλλάξουμε τα κοινωνικά κριτήρια» γιατί και εκείνες οι χώρες τελικά έχουν το βλέμμα στραμμένο προς εμάς και προσπαθούν ε, να ταυτιστούν με τις δικές μας ας πούμε κοινωνικές διαδικασίες. και βλέπουμε ότι ακόμα και σε μια κατάσταση όπως η τωρινή όπου οι πετρελαϊκές τιμές έχουν πέσει ε, ε, εξακολουθούν οι χώρες αυτές να ε, μπορούν να παραγάγουν πλούτο και επομένως καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά τα στοιχεία και να μην επικεντρωθούμε μονάχα στην πόλη στο πρώτο νηλόν. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριμένες και πιο εξειδικευμένες οι μέθοδοι αξιολόγησης. Εγώ ε, διαπιστώνω ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας αλλαγή στην ικανότητα αξιολόγησης. Αυτό μπορεί να πάρει χρόνο, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε περισσότερο και να κάνουμε πιο συγκεκριμένες ε, τι ε, μεθόδους αυτέ. και να επιμείνουμε σε την ε, αξιοπιστία των ίδιων των δωρητών. Μαζί με την Κομισιόν, στα πλαίσια μιας πολιτικής, ανταγωνιστική μιας συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων έχουμε λόγο ε, όσον αφορά αυτό το σημείο. Θα ήθελα επίσης ε, να δούμε τι θα κάνουμε ε, της fail state. Τι, τι κάνουμε δηλαδή στις χώρες οι οποίες δεν έχουν διακυβέρνηση. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό που θα μπορούσαμε τουλάχιστον να κάνουμε, και εδώ βέβαια θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των εταίρων χωρών, ε, να δούμε ποιος είναι ο χώρος ε, επί των οποίων μπορούμε να ε, αναπτύξουμε δράση με μη δημόσιους οργανισμούς, ας πούμε, με μη κυβερνητικές οργανώσεις. Η Επιτροπή μας υπέβαλε ένα ερώτημα και σε σχέση με την απάντηση θα ήθελα να υποβάλω εγώ το εξής ερώτημα. Τι θα γίνει, τι θα κάνουν τα, κράτη, τα Ηνωμένα Έθνη, τι θα γίνει ε, με την ε, ε, ανθρωπιστική βοήθεια στην Αντισαμπέμπα, τι θα κάνουμε με την πολυετή χρηματοδότηση, έτσι ώστε να σταματήσει αυτό το μπαλάκι που πετάει ο ένας τον άλλον είναι απαράδεκτη η κατάσταση αυτή. Δυσκολευόμαστε περισσότερο να πάμε να βρούμε το 5-10% που μένει παρά το να ε, μπορέσουμε να αντιλήσουμε ε, πόρους. Και νομίζω ότι θα πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Thank you, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο κύριος Σίλβα Περέιρα έκανε μια πάρα πολύ καλή αρχή της ε, συζήτησης σε σχέση με αυτό το, ε, την έκθεση ίδιας ε, πρωτοβουλίας και νομίζω ότι άνοιξε καλά το δρόμο για την Αντίσα Αμπέμπα όπου θα πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε παρόντες. Συμφωνώ, συμφωνώ απολύτως με το πρώτο σημείο το οποίο έθιξε σε σχέση με την δέσμευση. Εάν δεν δείξει την απαραίτητη δέσμευση η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε πώς περιμένουμε κάποιοι άλλοι να δεσμευτούν. Είχαμε υποβάλει χθε το ερώτημα ε, στην ε, Κομισιόν ε, για αυτές τις δεσμεύσεις. Μήπως δεν κατάλαβα καλά, αλλά έχω την εντύπωση ότι η Κομισιόν δεσμεύεται για το 0,7% σε σχέση με το τι θα κάνουν οι άλλοι. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό, ε, αυτός ο σωστός τρόπος. Ε, έχουμε απέναντί μας ε, αναπτυσσόμενες χώρες και επομένως ή θα δεσμευτούμε ή ας το αφήσουμε. Και ελπίζω αυτή να είναι η στάση και της Κομισιόν και των κρατών. Επίσης, η ανακοίνωση σε γενικές γραμμές είναι σχετικά καλά, καλή, περιλαμβάνει όλα τα ε, σωστά κεντρικά σημεία. Ε, θα θέλαμε βεβαίως να δούμε και μεγαλύτερη ε, δέσμευση όσον αφορά τον κατάλογο με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες πιστεύω και αναφέρθηκε από τους ε, συναδέλφους, ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες ε, θα έχουν την δυνατότητα ε, να πληρώσουν ένα κομμάτι της ανάπτυξης μόνοι τους μέσα από καλή διακυβέρνηση, ευφυείς πολιτικές, επιχειρηματικότητα κτλ. Αλλά για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες χρειάζεται αυτή η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Όσον αφορά την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, έχει εισαχθεί η νέα αρχή, η TOSD, δηλαδή ε, βοήθεια συγκεκριμένη για τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες, ε, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι θετικό γιατί επιτρέπει ευρύτερη κινητοποίηση πόρων για ευρύτερη ανάπτυξη. Ε, αλλά ελπίζουμε ότι πραγματικά θα αντικατοπτρίζει κάτι συγκεκριμένο και δεν θα εξαϊλωθεί ε, σε ε, έτσι, ασαφείς προτάσεις. Όσον αφορά την κινητοποίηση των πόρων, νομίζω ότι ο ΣΑ και ο πρόεδρος του είναι απολύτως δεσμευμένος, ε, ε, ο πρόεδρος Επιτροπής που είναι υπεύθυνος για τις αναπτυσσόμενες χώρες, είναι απολύτως δεσμευμένος ε, στα θέματα αυτά και έχει ξεκινήσει αυτό που ονομάζεται Tax Inspectors Without Borders, επιθεωρητές φόρων χωρίς σύνορα. Είναι μια πολύ καλή ιδέα. Συμφωνώ απολύτως με τους συναδέλφους που είπαν είναι σημαντικό να μπορούν να κινητοποιηθούν όλοι οι δυνατοί πόροι. Επίσης, αν μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα, πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε ότι ο ιδιωτικός τομέας θα, είναι, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Αλλά θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα παράδειγμα Ο πρώτος ε, ε, Υπουργός ε, Ανάπτυξης της Φιλανδίας κατάφερε να, λήξει το, το, Ταμείο Ανάπτυξης το οποίο τελικά δεν μπορούσε να βοηθήσει μέσω αυτών των υποτιθέμενων εγγυήσεων εξαγωγών πιστεύω ότι εδώ ελοχεύουν κίνδυνοι. Βλέπω ότι αυτό το εργαλείο ξαναέρχεται, επανακάμπτει. Ε, πολλές επικριτικές απόψεις είχα ακούσει για το ε, πόσο λίγο βοήθησε την ε, ανάπτυξη και πόσο λίγο ρόλο έπαιξε στην αναπτυξιακή βοήθεια. Ε, πρέπει να το προσέχουμε. Ε, ο εισηγητής ε, αναφέρθηκε επίσης ε, στις κατευθυντήριες γραμμές για συμπράξεις ιδιωτικού δημοσίου, πολύ σημαντικό. Ε, ε, για την διατύπωση αρχών ε, ορθής πολιτικής και ηθικής όσον αφορά την, το επιχειρήν. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα, αλλά δεν θα πρέπει να μας βγάζουν από το κεντρικό στόχο που είναι η, η χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Η διαφάνεια βεβαίως είναι ένα σημείο που ε, συζητιέται πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα πρέπει για μία ακόμα φορά ε, να υπογραμμίσουμε αυτήν την ανάγκη διαφάνειας και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά των δωρητών και από την πλευρά των αποδεκτών, ε, να είμαστε βέβαιοι δηλαδή με ποιους όρους δίνεται η βοήθεια και με ποιους όρους γίνεται δεκτή ότι φτάνει στον πραγματικό χρήστη. Τέλος, να υπενθυμίσω ότι θα έχουμε ε, και μία ειδική ε, έκθεση με εισηγητή τον κύριο Ντέβα όσον αφορά την ε, διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης. Πρόεδρος. Ναι, ε, βεβαίω υπάρχουν ε, πολύ ευρύτερα θέματα όπως είναι η φορολόγηση ή όπως είναι ε, άλλα ζητήματα συμπράξεων κτλ. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι τα, θέματα που θα ζητηθούν στην Αντίσα Μπέμπα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θέλω να επαναλάβω τα ίδια και τα ίδια. Να μην ξαναπώ αυτά που είπε η Χαουτάλα ο Σίλβα Περέιρα δούλεψε πολύ καλά. Παρόλα αυτά, παραμένει η δυσκολία προσέγγισης όσον αφορά αυτή τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη. Είναι γεγονός ότι έχουμε δωρήσει πολλά, ε, είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρώτος δωρητής, παρόλα αυτά υπάρχουν ε, μηχανισμοί οι οποίοι στην ουσία δεν έχουν ε, δημιουργήσει ανάπτυξη και συμμετοχικές διαδικασίες στις χώρες αυτές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να καταλάβουμε ποια είναι τα κατάλληλα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, γιατί αν από τη μία πλευρά μιλάμε για διευκολύνσεις ε, οι οποίες ενδεχομένως μπορεί να έχουν ε, ε, άσχημες επιπτώσεις. Από την άλλη πλευρά έχουμε το blending, την την ε, ανάμειξη δημοσίου και ε, ιδιωτικού χρήματος, αλλά που αν δεν αναμειχθεί σωστά τότε θα υπάρχουν προβλήματα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να αφήσουμε τα επιμέρους και να έχουμε μια ε, συνολική θεώρηση του τι συμβαίνει στον κόσμο. Μονάχα εάν έχουμε μια τέτοια ολιστική προσέγγιση θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τα πράγματα γιατί μπορεί να κάνουμε κάτι εδώ και να έχει ας πούμε επίπτωση στην κλιματική αλλαγή αλλαγή. Ε, ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι το σημείο κίνησής μας. σε γενικές ε, ε, γραμμές η έκθεση αυτή είναι καλή. Δεν ξέρω όμως αν θα έχουμε το χρόνο να συνεχίσουμε και στο μέλλον να δουλεύουμε με τον ίδιο ρυθμό. Δεν νομίζω ότι έχουμε τόσο πολύ χρόνο. Uh, thank you. Um... Ευχαριστώ πολύ. Με τη σειρά λοιπόν που φώναξα τα ονόματα, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή που παρουσίασε μια έκθεση η οποία είναι πολύ σημαντική. Πιστεύω πως θα είναι από τις μια πιο βασικές εκθέσεις ε, ιδίας πρωτοβουλίας φέτος και νομίζω ότι καλό θα ήταν να πέρασει εμπρόθεσμα από την Ολομέλεια έτσι ώστε να έχουμε και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου παράλληλα και όλα αυτά εν ώψη της διάσκεψης της Αντίσαμπέπα, έτσι ώστε να χαράξουμε την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διάσκεψη αυτή. Το ψήφισμα και η έκθεση θα στείλουν και ένα μήνυμα στους δικούς μας πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι σε πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζουν την χρηματοδότηση που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αναπτυξιακούς στόχους. Αναγνωρίζουν δε οι πολίτες μας ότι είμαστε μόνο το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού, είμαστε παράλληλα και το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Και είμαστε και το 50% της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Οπότε η διαφορά μεταξύ του 85% του παγκόσμιου ΑΕΠ με το 50% του παγκόσμιου, ε, της παγκόσμιας αναπτυξιακής ε, βοήθειας στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα για μια διεθνή σχέση όπου οι υπόλοιποι εταίροι θα έπρεπε να ανεβάσουν και αυτή τα ποσοστά χρηματοδότησης. Και νομίζω ότι θα πρέπει οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, να μάθουν πώς γίνεται αυτή η προσπάθεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να γνωστοποιήσουμε το μήνυμα αυτό στους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Όταν λοιπόν έχουμε ένα εσωτερικό θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ε, να δουλέψουμε στο εσωτερικό μας και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο έχει στείλει αυτό το ξεκάθαρο ε, μήνυμα πως χρειάζεται και πάλι να δεσμευθούμε στα πλαίσια μιας διεθνούς διαπραγμάτευσης έτσι ώστε να δούμε με ποιο τρόπο μπορούν οι υπόλοιποι ε, οι παγκόσμιοι εταίροι να ανεβάσουν τα δικά τους επίπεδα συνεισφοράς. Αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε κατά νου, στηρίζοντα προσπάθειες που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στι διεθνείς διαπραγματεύσεις. Χρειάζεται να ασκήσουμε κάποιες ε, πιέσεις έτσι ώστε να το πετύχει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σωστά ο εισηγητή αναγνώρισε τις τρεις πηγές, κάνα και μία ανταλλαγή απόψεων με τον εκπρόσωπο του ΩΣΑ και η σημασία της αναπτυξιακής βοήθειας φαίνεται να βαίνει μειούμενη, αλλά τοποθετήθηκε αυτό σε ένα διευρυμένο ε, περιβάλλον που πούμε ότι το 1% της αύξησης των φορολογικών εισόδων των αναπτυξιακών, των, ε, σε ανάπτυξη χωρών θα διπλασιάσει τη χρηματοδότηση τους ε, σε επίπεδα βοήθειας από το εξωτερικό. Αυτά λοιπόν εν ώψη της Αντισαμπέμπα και χαίρομαι που όσοι, όσα έχει τοποθετήσει ο σχόλια σε αυτή την έκθεση ο συγητής θα βοηθήσουν σημαντικά στην κατεύθυνση αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ θερμότατα τον εισηγητή για την περιεκτική παρουσίασή του και πραγματικά πιστεύω πως ανέφερε κάποια θέματα για την χρηματοδότηση και την έλλειψη δέσμευσης που πιστεύω πως είναι πάρα πολύ σημαντικά και πιστεύω πως ειδικά φέτος που είναι το Παγκοσμίο της Ανάπτυξης πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή για να τονίσουμε αυτήν την έλλειψη δέσμευσης και στο Νταβός και αλλού. Είναι ένα επιχείρημα το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Um, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Σίλβα Περέρη για την εξαίρετη εργασία του. Ευχαριστώ και τους ε, σκιώδεις για την πολύτιμη συμβολή τους. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω γιατί ε, και εκείνος και άλλοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν ε, στην δυνατότητα ε, κινητοποίησης των γηγενών πόρων. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθεί και αυτό ε, υπάρχει και άλλωστε αυτή η νέα έκθεση η οποία ε, θα ασχοληθεί με την φοροδιαφυγή ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες και θα γίνεται λόγος βεβαίως για την ανάγκη ύπαρξης σωστών, υγιών και ομοιογενοποιημένων φορολογικών συστημάτων και θα πρέπει βεβαίως να μιλήσουμε και για illicit financial flows είναι θέματα ε, στις χώρες αυτές ε, είναι θέματα τα οποία θα συζητηθούν ε, σε ένα σεμινάριο το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και οπωσδήποτε θα συνεχίσουμε τη συζήτηση και με την ευκαιρία αυτή της άλλης έκθεσης. Δεν βλέπω να ζητάει άλλος από τους συναδέλφους το λόγο. Θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποια σχόλια. Πριν δώσω το λόγο στην Κομισιόν και μετά στον εισηγητή, πιστεύω πως θα είναι μια εξαιρετικά σημαντική διάσκεψη και για το θέμα της αναπτυξιακής βοήθειας, όπως το είπε και ο συνάδελφος Ρούμπιχ, δεν σχετίζονται όλα με τα χρήματα. Έγινε μια παρουσίαση από τον Έρικ Σόλχαϊμ που είδαμε πως ε, τα χρήματα τα οποία είναι διαθέσιμα στα υποανάπτυξη κράτη είναι πολύ περισσότερο από αυτά που ε, προσφέρουμε εμείς με αναπτυξιακές βοήθειες. Δηλαδή 1% να αυξήσουν τους φόρους που συλλέγουν θα έχουν τα διπλάσια από όσα τους στέλνουμε εμείς αναπτυξιακή βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια στιγμή είπε πως οι διαπραγματεύσεις και στην Άντισα Μπέμπα και στη Νέα Υόρκη δεν θα σχετιστούν μόνο ε, με το θέμα αυτό, αλλά υπάρχει και μία στρατηγική παράταξη δυνάμεων γιατί θα εμφανιστούν η Κίνα ή οι αναδυόμενες ε, οικονομίες που θα προσπαθούν να παίξουν παιχνίδια εξουσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λοιπόν δεν επαναδεσμευτούμε για αυτό το ποσό, δεν θα μας ακούσουν καν στην υπόλοιπη συζήτηση. Θα μας πούνε πως η Δύση δεν είναι πρόθυμη να συζητήσει μαζί μας, άρα λοιπόν τους στρέφουμε την πλάτη. Άρα λοιπόν για να μας αφήσουν να μπούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα πρέπει εμείς να έχουμε και ένα αξιόπιστο χρονοδιάγραμμα και να δεσμεύσουμε αυτό το ποσό. Η αναπτυξιακή βοήθεια λοιπόν θα παίξει μεγαλύτερο ρόλο από ότι στην πραγματικότητα αξίζει γιατί θα είναι το κλειδί που θα μας φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και θα ακούσουμε και πάρα πολλά επιχειρήματα από τους εταίρους μας ε, για το τη φορολογία. Ναι, οι ε, αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να εξασφαλίσουν πως το φορολογικό του σύστημα φορολογικό σύστημα λειτουργεί. Και το επιχείρημα που θα μας, ε, με το οποίο θα μας απαντήσουν είναι ωραία. Και εσείς στη χώρα σας με το φορολογικό σύστημα είστε ικανοποιημένοι. Έχετε φοροδιαφυγή, έχετε φοροαποφυγή. Υπάρχει παγκόσμια συνεργασία έτσι ώστε να κατασταλούν αυτά τα φαινόμενα. Άρα λοιπόν όλοι πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά στο εσωτερικό μας για να καταφέρουμε να είμαστε έτοιμοι εκείνη τη στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα στοιχεία που έχετε από τον ΟΟΣΑ, πώς έχουν ληφθεί υπόψη στις δικές σας ε, εργασίες προετοιμασίας. Έχετε μια ειδική επιτροπή, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά έχει να κάνει με τα φορολογικά θέματα. Εκεί πώς λαμβάνετε υπόψη την εισφορά του όσα. Υπάρχει περίπτωση συμφωνίας σε επίπεδο ΩΣΑ που μπορεί να ερμηνευθεί ή να μεταφραστεί σε συμφωνία πριν την Αντισαμπέμπα από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στην ομάδα αυτή εργασία. Ματιέ Λεμό, σου δίνω το λόγο. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είσαστε λοιπόν εκπρόσωπος της DigiDevCo. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να αντιδράσουμε. Να σας πω πως καταρχήν καταγράφουμε όλα τα σχόλια τα οποία ακούστηκαν σήμερα και αναμένουμε το έτοιμο προϊόν. Πριν απαντήσω σε ερωτήσεις, θα ήθελα να κάνω κάποια πιο γενικά σχόλια. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για μας, το οποίο προσπαθήσαμε να περάσουμε μέσα στην ανακοίνωσή μας, είναι το θέμα της σφαιρικότητας. Δηλαδή, θα πρέπει η οπτική την οποία θα ακολουθήσουμε να είναι διευρυμένη σε σχέση με το παρελθόν. Όταν λέω λοιπόν σφαιρικότητα, μιλώ θα πρέπει να δούμε όλο το φάσμα των οικονομικών και μη οικονομικών ε, μνημονίων που έχουμε υπογράψει ε, έτσι ώστε να δούμε πώς θα εφαρμοστούν και να δούμε πώς θα κινητοποιηθούν οι εσωτερικοί πόροι, η πορεία από την αναπτυξιακή βοήθεια, τα διάφορα οικονομικά μέτρα και όλα αυτά να τα εξετάσουμε μαζί. Έχουμε το πρώτο σχέδιο για την Αντισαμπέμπα που είναι υποσυζήτηση στην ε, Νέα Υόρκη όπου μιλάμε ε, για την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο και το πώς θα βασιστεί αυτή στην αύξηση των εγχώριων πόρων. Επίσης, ε, τα χρήματα δεν μπορούν να αποτελέσουν τον πυρήνα των προσπαθειών μας. Θα πρέπει να είναι η καλή διακυβέρνηση αυτή η οποία θα στηρίξει την όλη προσπάθεια. Και βεβαίως έτσι επιστρέφουμε στο άλλο θέμα, στο θέμα των δεσμεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και έχουμε συνεισφέρει ιδιαίτερα σε όλους τους χώρους αυτούς. Μιλήσατε εσείς για το θέμα της ε, κινητοποίησης των εγχώριων πόρων. Εκεί στα πλαίσια της G20, των G20, κάναμε πολλή δουλειά και έχουμε διάφορα έργα εκεί, για παράδειγμα αυτόματη, αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών κατά της απάτης κτλ έτσι ώστε να διευρύνουμε και να πολλαπλασιάσουμε τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας που προσφέρουμε στα ε, αναπτυσσόμενα κράτη. Και μάλιστα ε, προτείνουμε ε, να εγκριθεί ως παγκόσμιο πρότυπο, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και το διαφορετικό δυναμικό που υπάρχει στα ευρωπαϊκά κράτη. Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η προσφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντως τέτοια είδους στοιχεία θα τα βάλουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στη διάσκεψη και γίνονται αυτή τη στιγμή συζητήσει και στο Συμβούλιο για το πώ θα ανταποκριθεί το Συμβούλιο στη δική μα ανακοίνωση. Εν πάση πτώση, αυτό είναι ένα κλάδο για τον οποίο πιστεύουμε πω έχουμε κάτι να φέρουμε στο τραπέζι. Για τι δεσμεύσει θα επανέλθω στο θέμα αυτό το απόγευμα και νομίζω θα σας τα παρουσιάσει ο Επίτροπος καλύτερα. Η έκθεση της γραμματείας του ΟΗΕ αποδεικνύει πως υπάρχει μια καλή ισορροπία μεταξύ των δεσμεύσεων και των μηνυμάτων που στέλνουμε και θα πρέπει να στηριχτούμε σε αυτό. Γνωρίζουμε πως ο κόσμος αλλάζει, ε, πως ε, θα πρέπει η ατζέντα και το πρόγραμμα που ακολουθούμε να είναι πιο παγκόσμιο εμβέλειας, το οποίο σημαίνει να μοιραστούμε τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και να προχωρήσουμε σε μια παγκόσμια εταιρική ε, σχέση. Αυτή η δέσμευση Ευρώπη συν 7 δεν θα πρέπει ε, να είναι δεσμευτική, θα την, θα την χαρακτηρίσουμε αναδέσμευση αν θέλετε ή εκ νέου δέσμευση, αλλά πρέπει να περάσει πρώτα από το Συμβούλιο. Χρειάζεται να σταθούμε όλοι με φιλόδοξο τρόπο και ίσως είναι λίγο νωρίς αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε σε μονομερείς κινήσεις σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να τοποθετηθεί στα πλαίσια ενός ευρύτερου πακέτου το οποίο θα συζητηθεί σε επίπεδο ΟΗΕ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής, κύριε Περέιρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλια. Θα κάνω μια πολύ σύντομη τελική παρέμβαση. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ξεκαθαρίσω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της ανακοίνωσής της έχει κάνει ένα πολύ θετικό βήμα στον χώρο της αναπτυξιακής βοήθειας και καλωσορίζω κάθε αναφορά που υπάρχει σε συνεκτικές πολιτικές, σε σφαιρική προσέγγιση. Είναι πολύ σημαντικά και στα οικονομικά μέσα εφαρμογής αλλά και για τα υπόλοιπα μέτρα τα εφαρμοστικά που προτείνονται. Αληθεύει πως χρειάζεται ε, επιμερισμός των ευθυνών και με τις νέες συνθήκες που ισχύουν στην παγκόσμια οικονομία αυτό έχει διαφορετική χρειά σήμερα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε όμως πως παρόλο που χρειάζεται να κινητοποιήσουμε επιπλέον και τους εγχώριους πόρους και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως η ιδιωτική χρηματοδότηση θα σταθεί δίπλα μας ε, στις προσπάθειες που γίνονται. Η δική μας βοήθεια παρόλα αυτά παραμένει σημαντική στα πλαίσια της αναπτυξιακής πολιτικής. Και αν θέλουμε στην να κάνουμε μια πραγματική γεμάτη νόημα συζήτηση για τα υπόλοιπα θέματα, δηλαδή ιδιωτική χρηματοδότηση, εγχώριους πόρους. Θα πρέπει να είμαστε απερίφραστα ξεκάθαροι στα θέματα τα οποία θα δείξουμε σε σχέση με την αναπτυξιακή βοήθεια. Διαφορετικά δεν θα το καταφέρουμε. Δηλαδή, νομίζω πως ε, μπορεί τελικά να κάνουμε ένα μεγάλο στρατηγικό λάθος. Να πάμε δηλαδή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να πούμε ναι, δεχόμαστε την έκκληση της Γραμματείας ε, των Ηνωμένων Εθνών για το 0,7%. Είμαστε έτοιμοι να σεβαστούμε και να ε, εκπληρώσουμε αυτό το στόχο. Υπό την προϋπόθεση πως οι υπόλοιποι ετάροι θα κάνουν το ίδιο και θα παρουσιάσουμε ένα χρονοδιάγραμμα. Υπό την προϋπόθεση πως οι εταίροι συμφωνήσουν με αυτό το χρονοδιάγραμμα και αν δεν παρουσιάσουμε καμία δική μας πρόταση και δεν την περιγράψουμε με κανένα τρόπο, τότε ε, η συζήτηση θα γυρίσει γύρω από το θέμα της αναπτυξιακής βοήθειας, την έλλειψη δεσμεύσεων, το πρόβλημα του χρονοδιαγράμματος και αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγάλος δωρητής αυτή τη στιγμή. Έχει ηγετικό ρόλο. Θα πρέπει λοιπόν να ηγηθούμε αυτή τη πολιτική συζήτηση στην Αντισαμπέβα και ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχουμε είναι εμείς να μιλήσουμε ξεκάθαρα για το ποιες είναι οι δικέ μας προτάσεις για την αναπτυξιακή βοήθεια. για να αποτελέσουμε υπόδειγμα για τους υπόλοιπους και νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να καταφέρουμε αυτά τα οποία επιδιώκουμε. Φοβάμαι πως δεν είναι μόνο θέμα τακτικής. Γιατί αυτή η ιδέα πως δεν θα παρουσιάσουμε εμείς χρονοδιάγραμμα γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμα εάν οι υπόλοιποι είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν τα δικά τους ε, συγκεκριμένους, δικούς τους συγκεκριμένους στόχους, μπορεί μεν να αποτελεί μία εξήγηση, αλλά υπάρχει άλλη εξήγηση. Να μας πούν πως το Συμβούλιο δεν συμφώνησε για το χρονοδιάγραμμα. Και ο πραγματικός λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παρουσιάζει χρονοδιάγραμμα είναι γιατί υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί, και υπάρχει μια σειρά χωρών που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο και δεν είναι έτοιμες αυτές οι χώρες ακόμα να αναλάβουν δεσμεύσεις. Άρα λοιπόν το πολιτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι αρκετά σύνθετο και δεν έχει να κάνει μόνο με την τακτική και τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε σε σχέση με τους υπόλοιπου εταίρους, αλλά έχει να κάνει και με τη δέσμευση που είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε ως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε δίκιο συνάδελφε, θα πρέπει να τονίσουμε και κάποια άλλα θέματα, εγχώριες, ε, πηγές εσόδων. Ε, ο Πολ Ρούμπιχ έχει δίκιο, θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να σταθούν στα πόδια τους οικοδόμηση δομών, επιχειρηματικό περιβάλλον, κράτος δικαίου, θεσμοί κτλ. Είναι πολύ σημαντικά. Αλλά αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο εάν παρουσιάσουμε μια συγκεκριμένη δέσμευση σε σχέση με την αναπτυξιακή βοήθεια, έτσι ώστε να δημιουργούν οι πολιτικές προϋποθέσεις ε, για να συζητήσουμε και όλα τα υπόλοιπα. Τέλος, την Γνάσιο σε διαβεβαιώνω πως όταν μιλάμε για διαφάνεια, λογοδοσία κτλ, Αυτό σημαίνει πως θα προχωρήσουμε και σε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Το λέει και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε σε μετρήσιμα απτά αποτελέσματα για να γνωρίζουμε αν η αναπτυξιακή μας βοήθεια πραγματικά πετυχαίνει κάποια αποτελέσματα. Και η διαφάνεια και η λογοδοσία περνάνε μέσα από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Με χαρά λοιπόν προσδοκώ να συνεργαστούμε έτσι ώστε να ετοιμάσουμε και το τελικό σχέδιο ε, πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά αρχίσαμε εξαιρετικά εδώ στην Επιτροπή. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία των σκιωδών εισηγητών. Να σας πενθυμίσω λοιπόν συνάδελφοι πως πρέπει να ψηφίσουμε την έκθεση στις 20 Απριλίου έτσι ώστε να είναι έτοιμη για την Ολομέλεια του Μαΐου και να εγκρίνουμε λοιπόν την έκθεση πριν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Προθεσμία για υποβολή τροπολογιών 23 Μαρτίου. Πότε θα μας στείλετε το κείμενο της έκθεσης, κύριε Περέιρα? Στο τέλος της εβδομάδας. Θα το στείλω για μετάφραση αυτή την εβδομάδα. Πολύ ωραία και θα το στείλουμε λοιπόν στους της συζητητής στα αγγλικά. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι η, η ακρόαση που θα γίνει σήμερα το απόγευμα με τον Επίτροπο Μίμητσα θα έχει επίσης καλεσμένους εκπρόσωπους μη κυβερνητικών οργανώσεων, εκπρόσωπους του ιδιωτικού τομέα και ε, του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτό το σημείο και ας προχωρήσουμε στο σημείο 11. Ελπίζω να είναι λιγότερο περίπλοκο το ζήτημα αυτό. Η Συμφωνία για το Εμπόριο, Ανάπτυξη και Συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ε, Νότιας Αφρικής προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ντάβορ Στύερ είναι ο εισηγητής. Του δίνω μέσο στο λόγο για να μας παρουσιάσει το θέμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι το θέμα αυτό είναι τεχνικό. Είναι ένα πρόσθετο πρωτόκολλο στην νομοθετική πράξη για την Συμφωνία Ρεμπόρια Ανάπτυξη και τη Συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νότιας Αφρικής. το πρόσθετο πρωτόκολλο προσθέτει την Κροατία ως νέο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος λοιπόν του πρωτοκόλλου αυτού είναι να ληφθεί υπόψη η Κροατία ως ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Να προσθεθεί η κροατική γλώσσα και υπάρχουν και κάποιες άλλες τροποποιήσεις τεχνικής φύσεως. Δεν υπάρχει κάτι επί της ουσίας για τη συμφωνία αυτή με την Νότια Αφρική. Η συμφωνία αυτή, να υπενθυμίσω ότι υπεγράφει το 1999 και τροποποιήθηκε το 2009 για να συμπεριληφθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας. Προς το παρόν, σε κάθε περίπτωση, έχουμε να κάνουμε με αυτό το πρόσθετο πρωτόκολλο που συμπεριλαμβάνει λοιπόν την Κροατία ως νέο μέλος της Ένωσης. Είναι μια τεχνική προσαρμογή. Το κείμενο θα σταλεί και μετάφραση αυτή την εβδομάδα. Υπάρχει 20 ε, Απριλίου ως ε, προσωρινή ημερομηνία ψηφοφορία στην Επιτροπή. Αλλά να σας πω ότι προς το παρόν αναμένουμε την απόφαση της ε, Νότιας Αφρικής όσον αφορά το ποιον θα εξουσιοδοτήσει για να υπογράψει τη συμφωνία. Υπάρχει επιθυμία από την πλευρά τους να υπογραφεί το κείμενο σε υψηλό επίπεδο, γι' αυτό λοιπόν ενδεχομένω να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση. Μετά πρέπει να σταλεί στο Κοινοβούλιο για έγκριση, το οποίο φυσικά μπορεί και να αρνηθεί αν θέλει, αλλά κάπως έτσι έχει το χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λίτς έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για την παρουσίαση αυτή. Όπως είπατε, είναι ένα τεχνικό ζήτημα. Η Νότια Αφρική είναι ένα στρατηγικό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένη τη επιρροή τη σε όλη την περιοχή τη Νότια Αφρικής. Βλέπουμε ότι η συμφωνία λειτουργεί πάρα πολύ καλά και συνδυάζει όλες τις πτυχές της με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Και φυσικά έχουν καλωσορίσει την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως έναν από τους ε, σημαντικότερους εταίρους. Όμως θα ήθελα εδώ να πάρω την ευκαιρία για να τονίσω τις προτεραιότητες που πρέπει να έχει η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής για να ολοκληρωθούν αυτές οι συζητήσεις διότι μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος ενδεχομένω υπονομεύσει την οικονομική κατάσταση όλης της περιοχής, την ανάπτυξη του εμπορίου στις ε, εκεί περιφέρειες και αυτό θα ήθελα να το αναφέρω για να δούμε λοιπόν τι θα κάνει η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής. Μάλιστα δεν βλέπω να θέλει κάποιος το λόγο, το Συμβούλιο θα ήθελε το λόγο. Υπάρχει κάποιος από την Γραμματεία του Συμβουλίου που θα ήθελε να μιλήσει. Όχι. Μάλιστα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν υπάρχει κανείς, αλλά κύριε Στήρα, έχετε να προσθέσετε κάτι. Όχι. Μάλιστα, ενημερωθήκαμε λοιπόν για το χρονοδιάγραμμα. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να το ψηφίσουμε τον Απρίλιο και ελπίζουμε να ψηφίσουν και οι Νοτιοφρικανοί. Περνάμε τώρα στο σημείο 12 συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την Συμφωνία TTIP. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων και σχέδιο γνωμοδότησης έγινε τον Ιανουάριο. Όπως ξέρετε, η Συμφωνία TTIP είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα δύσκολο και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη. Έχουμε 82 τροπολογίες στην γνωμοδότηση. Ελπίζω να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κάποιο συμβιβασμό σήμερα. Θα δώσω τώρα αμέσω το λόγο στον κύριο Λίτς, ο οποίος είναι ο εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία σας ε, στην εκπόνηση αυτής της γνωμοδότησης. Εμείς ε, πήραμε την απόφαση να είναι σύντομη, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες τροπολογίες ε, και βεβαίως προσπαθήσαμε να βρούμε συμβαστικό δρόμο. Προσπαθήσαμε να μην ε, προσπαθήσαμε και νομίζω ότι όλοι ακολούθησαν τη γραμμή να μην έχουμε ε, ε, πολύ, σημαντική, πολύ μεγάλη έκθεση. Έχουμε 7 συμβαστικές, ε, συμβαστικά σημεία, το ένα, το δύο, το οποίο ζητάει, ζητούσαν αρχικά οι σοσιαλιστικές και, οι σοσιαλιστικές και δημοκράτες, αλλά τώρα το ζητούν όλοι, νέους κανόνες για το TTIP. Τρίτον, συμβασμός ο οποίος αναφέρεται ε, στους κινδύνους του TTIP, συμβασμός 4 όσον αφορά τις ε, δεσμεύσεις. Ε, μετά ζητούμε με, την επόμενη, με τον επόμενο συμβιβασμό πολιτική δέσμευση, συμβασμός 6, ο οποίος ζητάει πολυμερείς συμφωνίες, οι οποίες, οι οποίες όμως συμπεριλαμβάνουν και τις διμερείς συμφωνίες και τελευταίο συμβασμός που αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και την πρόθεσή τους. Αναφερόταν ήδη στο προσχέδιο, αλλά θέλαμε πιο συγκεκριμένη αναφορά. Ε, και συμβασμός 8 που αναφέρεται στην, ε, στις οι οποίες δεν θα πρέπει να ε, υπάρχουν. Αυτά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Βεβαίως αν θέλετε σχόλια Λοιπόν, υπάρχουν 7 συμβιβαστικέ λύσει που έχουν προσυπογραφεί από όλε τι πολιτικέ ομάδε για να καταλάβουμε τι λέμε, λέει η Πρόεδρο. Ε, ωραία, έχουμε αυτού του συμβιβασμού λοιπόν που έχουν υπογραφεί από όλε τι πολιτικέ ομάδε. Ντάβοστ, πρώτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή Αναλίτσα για την εργασία του και για την προσπάθεια εξέβρεσης ε, συμβιβασμού ενώ ταυτόχρονα προσπάθησε να εστιαστεί στα ε, μηνύματα τα οποία θα πρέπει να στείλουμε μέσω ε, της γνωμοδότησης αυτής. Πιστεύω ότι οι συμβιβασμοί οι οποίοι έχουν βρεθεί όντως εκπροσωπούν τις διαφορετικές απόψεις Ε, βεβαίως υπήρχαν και κάποιες προτάσεις του ΕΛΚ που ε, μας δημιουργούσαν προβλήματα γιατί ήταν πολύ σκληρές γραμμές αλλά προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτή την επιπλέον προσπάθεια έτσι ώστε να βρούμε κοινό τόπο. Επίσης ε, και εμείς έχουμε, έχουμε αφαιρέσει, έχουμε βγάλει κάποιες τροπολογίες και εν πάση περιπτώσει αποφασίσαμε και να ε, ε, προσυπογράψουμε τον ε, συμβιβασμό που ανέφερε που είχαν υποβάλει οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες και που ανέφερε ο εισηγητής αποφασίσαμε να το στηρίξουμε έτσι ώστε να γίνει σαφές το θέμα της διαφάνειας επίσης αναφέρουμε στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων υπογραμμίζουμε και τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις του TTIP αυτό ήταν ήδη μια σημαντική δήλωση κατά την άποψή μας ευχαριστώ Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο Σάρλ δεν είναι εδώ. Σάρλ. Ε, Σάρλ Γκέρινγκ. Ε, έψαχνα μία τροπολογία. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι είναι η συμβαστική τροπολογία 8 που αφορά τη διαφάνεια της διαδικασίας όπου καλούμε την Κομισιόν να ε, ε, έχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Εδώ θα ήθελα να πω καλούμε την Κομισιόν και το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη. Ε, ε, θέλω να κάνω αυτή την προφορική τροπολογία γιατί ε, τα κράτη-μέλη αποφασίζουν εάν η εντολή θα είναι δημόσια ή όχι. Δηλαδή θα πρέπει όχι μόνο να ζητήσουμε την Κομισιόν αλλά να είμαστε βέβαιοι ότι δέχονται αυτήν την δημόσια ανοιχτή διάφανη εντολή τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό ζητώ την έγκρισή σας. Ναι, ε, λέει η Πρόεδρος, κάνετε μία προφορική τροπολογία για το συμβιβασμό 8, αλλά δεν υπάρχει ο συμβιβασμός 8. Ναι, συμβιβασμός 8 που λέει καλεί την Κομισιόν ε, να δημοσιοποιήσει περισσότερα έγγραφα ε, διαπραγμάτευσης. Ναι, αλλά ε, ε, για να δημοσιοποιηθούν τα έγγραφα θα πρέπει αυτό να γίνει ε, όχι μόνη της, δεν μπορεί να το κάνει συγγνώμη μόνη της η Επιτροπή, αυτό πρέπει να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη των, και την άδεια των κρατών μελών. Εντάξει, θα επανέλθει μετά στο τέλος ο, ο εισηγητής, γιατί είχα την αίσθηση ότι ο, ο συμβασμός 8 δεν υπάρχει πια. άλλα Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ο Σλένφος Λίτζε πραγματικά συνεργαστήκε με όλες τις πολιτικές ομάδες και πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμη η συμβιβασμοί. Και υπό το φως και της τελικής έκθεσης της Επιτροπής Ίντα. Το μόνο πρόβλημα το οποίο εξακολουθούμε να έχουμε είναι ο συμβασμό 4, γιατί κατά την άποψή μας είναι εξαιρετικά αισιόδοξο όσον αφορά ε, την δυνατότητα οι συμφωνίες TTIP και IP να δημιουργήσουν πραγματικά ένα ε, καλό αποτέλεσμα σε καλή συνεργασία. Ενδεχομένως να υπάρξουν ευκαιρίες, αλλά σίγουρα δεν είναι μόνο ευκαιρίες αυτές που θα παραχθούν από τις ε, συμφωνίες. Θα ήθελα λοιπόν να δείξουν ευελιξία οι συνάδελφοι έτσι ώστε ε, να προσεγγίσουν την κατά την άποψή μας πιο ισορροπημένη ε, διατύπωση. Κατά τα λοιπά, συμβιβασμός 8. Δεν νομίζω ότι η Επιτροπή Ανάπτυξης ε, είναι η κατάλληλη για να κάνει λόγο για την ε, ε, διαφάνεια. Ε, ίσως άλλες επιτροπές να είναι πιο αρμόδιες, να το αφήναμε λοιπόν για τις άλλες επιτροπές. Δεν ξέρω. Όσον αφορά τώρα την παρατήρηση του Σαλ για την πρόσβαση στα έγγραφα. Δεν νομίζω ότι ισχύει πραγματικά και πλήρως το ότι η Κομισιόν μόνη της δεν μπορεί να δημοσιοποιήσει έγγραφα γιατί ο, ε, ο σχετικός κανονισμός προβλέπει κάποιες ε, εξαιρέσεις. Νομίζω ότι έχει δυνατότητα και η Κομισιόν. Δεν ξέρω, ίσως υπάρχει μια σχετική σύγχυση εδώ. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα της διαφάνειας όντως είναι κεντρικό σημείο, απλώς δεν είμαι βεβαία ότι η Επιτροπή μας είναι το κατάλληλο φόρουμ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανελής. Θα ξανασυζητήσουμε τα προβλήματα αυτά ε, στο μέλλον ο Ιγνάτσιο μετά και μετά ο Σάλς. Ιγνάτσιο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Λίτς για την εργασία που έχει κάνει. Βέβαια έγινε ακουστή η φωνή όλων, ήταν πράγματι ε, πολύ συνολική δουλειά και αυτό είναι πολύ κακό. Καλό, συγγνώμη όσον αφορά το TTIP, νομίζω ότι ε, είναι κακή η συγκυρία στην οποία δημιουργήθηκε, ε, κακή η μοίρα κατά από την οποία δημιουργήθηκε αυτή η συμφωνία και νομίζω ότι αυτό διαφαίνεται και από τις ε, συζητήσεις της άλλης Επιτροπές. Βεβαίως εμείς εξετάζουμε τις επιπτώσεις που θα έχει η συμφωνία αυτή στις αναπτυσσόμενες χώρες και ε, συμφωνώ με τη συνάδελφο ότι το να έχουμε ένα τόσο ευχάριστο και αισιόδοξο τόνο στο συμβασμό 4 είναι υπερβολικό. Θα ήμουν εγώ πάρα πολύ προσεκτικός όσον αφορά τη διαφάνεια για το κατά πόσον είναι αρμοδιότητα δικιά μας της Επιτροπής μας να μιλάμε για τη διαφάνεια. Εγώ πιστεύω ότι η διαφάνεια είναι μια απόλυτη αξία, μια απόλυτη αρχή η οποία θα πρέπει πάντα και με κάθε τρόπο να επιδιώκεται διαφάνεια στη διαπραγματεύση, σε διαφάνεια ε, στα στοιχεία της ε, ε, συμφωνίας αυτής. Και η έλλειψη διαφάνειας βέβαια ήδη σηματοδοτεί κάποια στοιχεία για την συμφωνία αυτή. Πάντως θα ήθελα για μία ακόμα φορά να συγχαρώ τον συνάδελφο και να τον ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία και τη δυνατότητα που έδεσε σε όλους να ακουστεί η φωνή τους. Λάουρα Σάντσα, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν του συνάδελφου για τη δουλειά που έκανε. Έχω κάποια σχόλια όμως. Καταρχήν απευθύνω μία έκκληση σας, συνάδελφοι. Θα ήθελα να στηρίξετε την τροπολογία 76 έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε επισήμω ε, και τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη της ε, κοινωνίας των πολιτών. Γιατί η άλλη τροπολογία που απλώς ζητά την πρόθεση του διαλόγου με την ε, κοινωνία των πολιτών δεν επαρκεί. Και σε σχέση με τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την TTIP και την διαφάνεια, τότε να τη ζητήσουμε να προωθήσει ε, τον διάλογο. Αλλά η απλή προώθηση, τι να σας πω, είναι κενό γράμμα, γιατί αν ζητά πραγματικά διαφάνεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι γιατί το απαιτεί η κοινωνία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αναφέρεται με δεσμευτικό τρόπο. Χτες ε, στην Μαδρίτη εγώ συζήτησα ε, με τον επικεφαλής των διαπραγματεύσεων και είναι ξεκάθαρο, είναι η κοινωνία των πολιτών που πιέζει και που αναγκάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει τη διαφάνεια. Συμφωνώ με τον Ιγνάσιο Είναι εγκάρσιο θέμα της δημοκρατίας η διαφάνεια. Αν δεν έχουμε διαφάνεια δεν υπάρχει δημοκρατία. Άρα λοιπόν όλες οι επιτροπές θα πρέπει να ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πιο διάφανη στις εργασίες της. Για την τροπολογία 80 που απευθύνει μία έκκληση να είναι ε, προσβάσιμα όλα τα έγγραφα, πρέπει να σας πω το εξής. Η διαφάνεια την οποία επικαλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πραγματικότητα δεν σημαίνει τίποτα. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε τα ε, ολοκληρωμένα ε, κείμενα, τα τελικά κείμενα, τα οποία είναι αδύνατο να δούμε και μας λένε δεν γίνεται γιατί θα αποκαλύψουμε τη στρατηγική των διαπραγματεύσεων. Ναι, αλλά τα συμφωνημένα κείμενα δεν εμπίπτουν σε αυτή την ε, ε κατηγορία. Καταπίπτεται αυτό το επιχείρημα γιατί τα παγιωμένα ε, τελικά κείμενα τα έχουν δει και οι δύο πλευρές. Άρα λοιπόν εμάς γιατί δεν μας τα δείχνετε. Αυτό μας ενδιαφέρει. Γιατί, και το λέω για τη θέση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό το οποίο τελικά έχουμε στο τελικό κείμενο είναι κοντά στις προτάσεις αρχικής της Κομισιόν ή είναι κάτι που είναι αρκετά μακριά. Θέλουμε να το δούμε γραμμένο στο χαρτί και να σας πω πως υπάρχει και απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ζητά περισσότερη διαφάνεια και ζητά να μην χρησιμοποιείται σε εξαίρεση τον κανονισμό αυτό για την διατήρηση του απορρίτου ως γενικό κανόνα, όπως κάνει μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, να, να ε, χρησιμοποιείται ως εξαίρεση. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό το σημείο αυτό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να απαιτήσουμε εμείς όλες οι επιτροπές να έχει μεγαλύτερη διαφάνεια, γιατί χωρίς διαφάνεια δεν θα έχουμε δημοκρατία. Αυτό ήταν το σχόλιο μου. Thank you. Charles, you want to say something else? Charles, θέλεις να κάνεις και εσύ κάποιο σχόλιο. Ναι, θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ σε μια προφορική τροπολογία την οποία έχω καταθέσει και να προσθέσω και τα κράτη-μέλη and the member states. Και σας λέω γιατί. Εγώ αναφέρθηκα στην δημοσίευση της εντολής. Η εντολή ορίζεται από τα κράτη-μέλη και ε, παραδίδεται στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκτέλεση αυτής της εντολής. Αλλά όσο το τελευταίο κράτος μέλος που ε, δεν ήθελε να δημοσιευθεί αυτή η απάντηση, όσο δηλαδή υπάρχει άρνηση έστω και ένα κράτος μέλος, δεν μπορεί να δημοσιεύσει την εντολή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και γι' αυτό πρότεινα να εισάγουμε αυτή την τροπολογία. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο στα όσα είπατε. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι υπάρχει διαφάνεια για το Κοινοβούλιο. Η ευθύνη λοιπόν της διαφάνειας καλύπτει με τον πιο δευρυμένο τρόπο που γίνεται το Συμβουλίο, τα κράτη-μέλη και βέβαια κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αν υπάρχουν αμφιβολίες μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με την νομική υπηρεσία για να μας εξηγήσει τι γίνεται. Χέιτι, όχι για το σημείο αυτό. Καταρχήν στηρίζω απόλυτα αυτή την προσθήκη, δηλαδή και τα κράτη-μέλη να δημοσιεύουν την εντολή όταν εγκριθεί. Ένα μισό χρόνο πήρε. Και τελικά μόνο επειδή υπήρξε πάρα πολύ πίεση τα καταφέραμε. Έχουμε άλλη μία, άλλο ένα παράδειγμα τώρα. Η Επίτροπος Μάλστρομο έχει ζητήσει, παρακαλέσει, απευθύνει έκκληση ε, για να δημοσιεύσουν την εντολή για τις υπηρεσίες ε, τα κράτη-μέλη. Θέλουμε λοιπόν μια αλλαγή κουλτούρας, σύμφωνα με τα όσα είπε και η συνοδελφός μας, έτσι ώστε να ενεργοποιείται αυτό αυτόματα. Νομίζω πως είναι πολύ σύνθετο το θέμα και για τη δημόσια πρόσβαση αλλά και για τα δικά μας δικαιώματα ε, αυξημένης ε, πρόσβασης. Αυτή τη στιγμή αναμένεται μία μελέτη από τους εμπειρογνώμονες τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δει τα δύο θέματα αυτά. Και στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συζητήσαμε σήμερα το πρωί πως θα περιμένουμε να κατατεθεί η μελέτη έτσι ώστε να εστιάσουμε στο πώς θα πρέπει το Κοινοβούλιο να ενημερώνεται λαμβάνοντας υπόψη την συνθήκη της Λισαβόνας όπου ε, ακόμα και σε συμφωνίες τύπου TTIP το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει ή όχι. Ποια είναι η σωστή στιγμή της ενημέρωσης είναι το ερώτημα κλείδι για μας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι καταλήγουμε σε μία μάλλον χλιαρή λίστα απαιτήσεων για την διαφάνεια. Εδώ χρειάζεται κάποια πίεση από πλευράς κοινοβουλίου. Ξέρω ότι κάποιοι ασχολούμαστε πολύ με το θέμα. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρουμε. Να ρωτήσουμε τον Άρνη, γιατί ο Σαλ έχει υποβάλει τροπολογία για ένα συμβιβασμό που δεν υπάρχει, θέλει να τροποποιήσει και κάτι άλλο παράλληλα. Δεν μπορούμε και δεν χρειάζεται να τα λύσουμε όλα σήμερα για τη διαφάνεια. Είναι τεράστιο το θέμα και είναι μεγάλο θέμα για ολόκληρο το Κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν είναι γνωμοδότηση προς την ίντα και θα πρέπει να ενταχθεί στα κείμενα της ίντα. Οπότε ίσως η ίντα ζήτησε τη μελέτη ακριβώς γιατί είναι τόσο περίπλοκο. Οπότε εμείς δεν χρειάζεται να λύσουμε τα ζητήματα αυτά σήμερα εδώ. Και δεν θα έχουμε και την τελική... Δεν θα πούμε εμείς την τελική λέξη γιατί είναι μια πρώτη γνωμοδότηση, θα συντονιστούμε, θα μελετήσουμε, θα δούμε και τις επιπτώσεις ε, στα αναπτυξιακά θέματα της TTIP, αλλά μόνο όταν έχουμε περισσότερα στοιχεία για την TTIP θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα για το ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της και θα πρέπει να γνωρίζουμε τις παραμέτρους αυτής της συμφωνίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε το λόγο, με συγχωρείτε, ο κύριος Μπουρσιέ από την Γενική Διεύθυνση Trade. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για το ζήτημα της TTIP και το πώς επηρεάζει την ανάπτυξη. Να σας πω καταρχήν πως όντως υπάρχει αυτή η διάσταση. Υπάρχει υποχρέωση της ε, συνθήκης να εξασφαλίσουμε πως υπάρχει συνέπεια μεταξύ της πολιτικής για την ανάπτυξη και των υπολείπων. Υποβάλλουμε τακτικές εκθέσεις και στην επόμενη έκθεση για τις επιπτώσεις της TTIP στην ανάπτυξη θα ληφθούν τα στοιχεία δεόντως υπόψη. Φυσικά, γνωρίζοντας το βάρος που έχουν η ευρωπαϊκή και η αμερικανική οικονομία και το τι σημαίνουν οι ευρωπαϊκές και οι αμερικανικές αγορές για τις χώρες τις αναπτυσσόμενες, τα όσα θα συμβούν μεταξύ των δικών μας αγορών εν δυνάμει ε, έχουν σημαντικές επιπτώσεις για τις τρίτες χώρες, για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Να πω απλώς πως το θέμα αυτό ήδη σε κάποιο βαθμό έχει εξεταστεί σε μία μελέτη που, που ζήτησε η Κομισιόν <coughs> από το Κέντρο για, το... για τις Έρευνες Οικονομικής Πολιτικής το οποίο είχε καταλήξει πως θα είναι θετικές οι συνέπειες για τις τρίτες χώρες από τη Συμφωνία TTIP και κυρίως για τις χώρες με χαμηλά εισοδήματα. Αλλά δεν περιορίζεται σε αυτές. Το ζήτημα θα αναλυθεί με λεπτομέρειες στα πλαίσια της έκθεσης ε, επιπτώσεων στη βιωσιμότητα που τρέχει παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις. Και ο τρόπος με τον οποίο εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζουμε τα θέματα αυτά είναι ο εξής. Υπάρχουν δύο διαφορετικές διαστάσεις υπάρχει η παραδοσιακή ανταλλαγή, ε, εμπορική ανταλλαγή και υπάρχουν και κάποια κανονιστικά θέματα τα οποία συνδέονται με την ε, σχετική συμφωνία με τις είπα για το θέμα αυτό, για την παραδοσιακή διάσταση, δηλαδή τις εμπορικές πτυχές και συνέπειες. Το εμπόριο όντως ε, παραδοσιακά αυξάνει το ΕΠ και στη ΣΥΠΑ και στην Ευρώπη. Πάνω από 120 δις θα αυξήσει το ΕΠ στην ε, Ευρώπη λόγω της ε, διόγκωσης της, ε, των συναλλαγών στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό θα ωφελήσει και τις τρίτες χώρες. Τώρα, για τις τρίτες χώρες, το τι θα γίνει με, την εμπορική, με τις εμπορικές ρυθμίσεις και το τι θα γίνει σε επίπεδο ανταγωνισμού με τους με τις χώρες που μας εφοδιάζουν εμάς και την Αμερικανική αγορά, εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ενδεχομένως, σε κάποιες συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις μπορεί να έχουμε επιπτώσεις. Αλλά αν δούμε σε γενικές γραμμές τις πιο αδύναμες χώρες και τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, αφρικές χώρες, αφρικανικές χώρες για παράδειγμα, δηλαδή αναλόγως με το ποια ομάδα θα επιλέξουμε, αν δούμε λοιπόν τα 10 βασικά αγωθά εξαγωγής ε, εξαγωγικά αγαθά των λιγότερων αναπτυσσόμενων χωρών που είναι από το 70 μέχρι το 80% των εξαγωγών τους, κανένα δεν έχει τίποτα κοινό με τα 10 βασικά εξαγωγικά προϊόντα των ΗΠΑ προς την Ευρώπη και αντίστροφα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης, οι λιγότερες ανεπτυγμένες ε, χώρες ε, που εξάγουν στην Ευρώπη εξάγουν τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που μας εξάγουν οι Ηνωμένε Πολιτείες. Αυτό είναι λοιπόν ένα στοιχείο που συνδέεται με αυτές τις κλασικές συμφωνίες ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών. Το δεύτερο θέμα είναι συγκεκριμένα το κανονιστικό πλαίσιο. Και στις συζητήσεις που γίνονται για τις επιπτώσεις στην TTIP και στην ανάπτυξη γίνεται μία συζήτηση για τους φραγμούς ε, στην είσοδο των προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά που ενδεχομένως θα έρθουν οι υγειονομικά και φυτογειονομικά προϊόντα. Δεν είναι ξεκάθαρο πως τα όσα γίνονται στα πλαίσια της TTIP σε κανονιστικό επίπεδο TBT, SPS κτλ. δεν θα επηρεάσουν καθόλου με την άρση των φραγμών. Θα διευκολύνουν τις συναλλαγές όπου γίνεται αλλά δεν σημαίνει πως θα άρουν φράγματα είτε από τις, μεταξύ ΙΠΑ Ευρώπης είτε μεταξύ τριών, τρίτων χωρών και ΙΠΑ Ευρώπης. Βεβαίως υπάρχει ένας ε, συντονισμένος τρόπος, ε, μάλλον όχι συντονισμένος, αλλά ένας ε, διάλογος στη στιγμή που επιβάλλουμε κανονιστικές διατάξεις από όλες τις διώχθες του Ατλαντικού. Αυτό θα έχει και θετικές επιπτώσεις για τι τρίτε χώρε γιατί θα είναι πιο διάφανη η νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή, στην ε, πιο διάφανη σχετική νομοθεσία και αυτό είναι θετικό, περισσότερο παρά Υπάρχει και ένα κάθετο ε, κλαδικό θέμα για τη συνεργασία κάποιων ε, κλάδων μεταξύ τους. Εκεί ο στόχος είναι η ευρωπαϊκή προσέγγιση, η αμερικανική προσέγγιση να είναι παρόμοια με μια αξιολόγηση κινδύνου, για παράδειγμα για τα αυτοκίνητα οχήματα να είναι κοινή, απαρόμοια και να αναγνωρίζετε πως υπάρχει ισοδυναμία μεταξύ των προσεγγίσεων που υπάρχουν έτσι ώστε να διευκολύνουμε τους εμπορικούς φορείς. Αντί να χρειάζεται δύο φορές να καλύψουν δύο διαφορετικά σετ συγκεκριμένων απαιτήσεων ε, από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι υπάρχει αρνητική επίπτωση από αυτό για τι τρίτε χώρε, μάλλον θετική είναι γιατί θα μπορούσαν ε, και ε, σύντο χρόνο να συμμετέχουν και αυτές σε αυτό το μηχανισμό. Και τέλος, η σχέση με τον ΠΟΕ, έχουμε μία παράγραφο στο σχέδιο γνωμοδότησης για το συγκεκριμένο θέμα και πρέπει να σας πω πως εγώ μάλλον το χρωματίζω κάπως παραπάνω γιατί από τη στιγμή που θα συμφωνήσουν για κάποια θέματα είπα Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολυμερές επίπεδο δεν υπάρχει αυτοματοποίηση των ε, εισαγωγών. Όχι. Το μόνο που υπάρχει είναι μια συνεισφορά τον ΙΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πολυμερή συζήτηση. Δυστυχώς οι πολυμερές διαπραγματεύσει έχουν ε, διακοπή λόγω κάποιων εμπλοκών και καλό θα ήταν ε, κάποιες συζητήσεις εκεί να ξαναξεκινήσουν και αν ε, κινηθούν οι ΙΠΑ και αναλάβουν πρωτοβουλία και δείξουν τη διάθεση ηγεσία, θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε φραγμούς που δημιουργεί διαφορετική παράδοση μεταξύ ΙΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και ίσως θα επιτρέψει αυτό στο πολυμερές σύστημα να προοδεύσει και αυτό κάπως πιο γρήγορα ε, στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος. Και τέλος για τη διαφάνεια που συζητήθηκε προηγουμένως, να σας υπενθυμίσω πως αποτελεί προτεραιότητα της ε, Επιτρόπου Μάλστρομ από τη στιγμή που ανέλαβε τη θέση αυτή και νομίζω ότι υπάρχει πραγματική αναγνώριση και ευαισθητοποίηση του πόσο σημαντική είναι η διαφάνεια για τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις και για όλα τα κανονιστικά θέματα που έχουν ε, δημιουργήσει ερωτηματικά και συζητήσει στην Ευρώπη, υπάρχει μια ευαισθητοποίηση και υπάρχει η πρόθεση συζήτησης, πρόοδου, γιατί πρέπει να σου πω ότι αντικειμενικά δεν ήμασταν ποτέ τόσο διάφανοι στις διαπραγματεύσεις που κάνουμε σε διμερές επίπεδο. Η εντολή διαπραγμάτευσης τελικά δημοσιεύθηκε, πολύ καθυστερημένα, το ξέρετε. Η θέση της Κομισιόν από την αρχή ήταν πως πρέπει να δημοσιευθεί. Και πέραν αυτού υπάρχει μεγάλη όρεξη από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κάνει ό,τι μπορεί η ίδια σε επίπεδο δημοσίευσης κειμένων ε, τα οποία η ίδια καταθέτει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και να σας πω ότι αρχές Ιανουαρίου, πριν από ένα μήνα δηλαδή περίπου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα περισσότερα κείμενα που παρουσίασε ως διαπραγματευτικά κείμενα και για τα κανονιστικά θέματα ε, αυτά αποτελούν πια και αυτό αντικείμενα δημόσια συζήτησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Για να διευκρινίσω κάτι. Ε, αναφέρθηκε μια μελέτη για, την, ε, για τις επιπτώσεις σε τρίτες χώρες από την Επίτροπο Μάλιμστρομ. Αν δεν κάνω λάθος, πότε θα την έχουμε αυτή την έκθεση. Όχι, αυτή η μελέτη, μια μελέτη ε, η ΣΕΠΑ, είχε δημοσιευθεί πριν από δύο χρόνια και είχε συμπεριλάβει και τη διάσταση τρίτων χωρών. Στα πλαίσια της ε, εκτίμησης αντικτύπου για τη βιωσιμότητα, στις ε, τρίτες χώρες και είχαν συμπεριληφθεί και χώρες με χαμηλό εισόδημα. Στην ε, συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο Σούλτς αναφέρθηκε μία μελέτη για τις τρίτες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν θα μπορούσατε να μας ε, δώσετε περισσότερες διευκρινήσεις έτσι ώστε να μάθουμε περισσότερα. Γιατί αυτό μας είπε η Επίτροπος Μάλμστρομ στο Στρασβούργο. Και αυτό έχει συζητηθεί και με τον πρόεδρο Σούλτ. Ε, κύριε Γκέρντ, είναι πηγών. Μία ερώτηση στην Κομισιόν. Αυτή, ε, ε, ε, αυτό που ανέφερε όσον αφορά τον αντίκτυπο της, για τη βιωσιμότητα, τι θα γίνει. Υπάρχει, υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι χώρες ΑΚΕ, οι οποίες όμως σιγά σιγά αναπτύσσουν, αναπτύσσονται, άρα φεύγουν από τις λιγότερο αναπτυγμένες ενδεχομένως μπορούμε να βοηθήσουμε ε, τις ε, ε, χώρες μέσω τεχνογνωσίας έτσι ώστε να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους. Αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο απλό. Νομίζω πως ήδη είχαμε μια απάντηση γι' αυτό, αλλά ας περιμένουμε τη μελέτη. Γιατί νομίζω πως τα δικά μας πρότυπα έτσι κι αλλιώς είναι υψηλότερα από τα Αμερικανών, οπότε ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη μελέτη. Έτσι κι τα πρότυπα στι ΗΠΑ μπορεί να αλλάξουν. Αλλά σας παρακαλώ ε, αφήστε να δώσω το λόγο στον κύριο Λίτς για να τελειώσει. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, πολλέ τοποθετήσει σα. Θα ήθελα να πω ότι με εξέπληξε η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι η Επίτροπος είχε ανακοινώσει αυτά τα πράγματα, μας είχε πει ποτέ θα δημοσιευτεί αυτή η μελέτη. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε περισσότερες πληροφορίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή και για αυτή την γνωμοδότηση. Και στην Γερμανία να σας πω ότι το Κοινοβούλιο έχει δώσει την εντολή να γίνουν πάρα πολλές μελέτες, όμως εδώ δεν έχουμε μία επαρκή βάση έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, να συντάξουμε δηλαδή αυτή τη γνωμοδότηση. Τώρα, η ε, κυρία Χάουταλε για τις ε, συμβαστικές λύσεις 3 και 4 σχετίζονται μεταξύ τους αυτές οι δύο συμβαστικές προτάσεις. Επίσης, και ο κύριος Σάντσες, αν δεν κάνω λάθος, είπε κάτι για ένα ενοποιημένο κείμενο. Πιστεύω πως είναι μια καλή προσέγγιση, πολύ ενδιαφέρουσα και θα μπορούσαμε να την ακολουθήσουμε ή να βάλουμε να προσθέσουμε κάτι εκεί για το πότε θα πρέπει να δημοσιευθεί κάτι και πρέπει φυσικά να έχουμε την έγκριση των εθνικών κοινοβουλίων. Βέβαια φυσικά και κατανοώ τις ανησυχίες σας περί διαφάνειας, όμως ε, άλλο συζητάμε τώρα να βρούμε ένα συμβιβασμό. Κύριε Κέρεντς, Θα σας απαντήσω γραπτά. Ναι, και τα κράτη-μέλη. Αυτό ήθελα να πω, τίποτα παραπάνω, να προσθεθεί. Λοιπόν, τότε νομίζω πως ε, πρέπει να συναντηθούμε όλοι οι σκιώδεις εισηγητές, ίσως και σήμερα το απόγευμα και όλες. Και αν είναι έτσι όπως μου τα λέτε, τότε θα προτείνω να διαγραφεί 81 αλλά δεν μπορώ να σας πω αμέσως, πρέπει να το κοιτάξω. Αυτά τα λίγα από μένα. Μάλιστα, θα σας αφήσω λοιπόν κύριε Λίτς να τα βρείτε με τον κύριο Γκόρεντς σήμερα το απόγευμα. Θα μπορούσε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας διευκρινίσει το θέμα αυτό με τη μελέτη. Είναι επίγον και σας παρακαλώ κιόλας να είστε λίγο σύντομος αν μπορείτε. Λοιπόν, να ενημερώσω ότι η ψηφοφορία για τη γνωμοδότηση θα λάβει χώρα σήμερα το απόγευμα. Έχουμε συμβιβαστικέ τροπολογίε, οπότε ελπίζω να τελειώσουμε γρήγορα με την ψηφοφορία. Και πιστεύω πως αφού δούμε τη νέα μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και θα ξέρουμε περισσότερα. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.